Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι ξενούμενοι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την ημερήσια διάταξη. Εν τω μεταξύ, οι διερμηνείς θα ήθελαν να κάνουν μια ανακοίνωση. Βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα κινητοποιήσεων λόγω τη εργασιακή διάνεξη με τη διοίκηση για τι συνθήκε εργασία. Σε ορισμένε καμπίνε έχουν επιστρατευτεί όλοι οι διερμηνείς και είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν. Αυτό καταργεί το δικαίωμά του στην απεργία και συνιστά διάκριση. Η ελληνική καμπίνα δεν θα προχωρήσει σε στάση εργασία που προβλεπόταν για τη σημερινή συνεδρίαση. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ε, το θέμα το οποίο μα απασχολεί εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε η Ήπειρος η οποία ε, καλύτερα προστατεύει τα προσωπικά ε, δεδομένα, αλλά είμαστε ε, η, η η οποία λιγότερο προστατεύει τα πολιτιστικά δεδομένα και αυτό είναι ανεξήγητο. Επομένως, κύριε Πρόεδρε, χρειάζεται μεγάλη ηρεμία στην ψηφοφορία την οποία θα κάνουμε σήμερα και την οποία παρακολουθούν πολλοί κόσμος, πολίτες της Ευρωπαϊκής Υπήρου, εκπρόσωποι του σχετικού κλάδου, ε, όλοι δηλαδή όσοι ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ ε, για κάτι το οποίο ε, ούτε προηγούμενο έχει, ούτε αποδεκτό είναι. Μαθαίνω ότι μας πίεσαν ε, προσπαθώντας πρώτα να μας υποχρεώσουν ε, για να ψηφίσουμε πρώτα από το κείμενο τα, τις προφορικές αυτό δεν είναι αποδεκτό. Δεύτερον και πιο σημαντικό, με μια παθητικότητα για να μην πω στην ενοχή της γραμματείας και το λέω με τα λόγου γνώσεως, μα υποχρεώνουν να ψηφίσουμε τις αιτιολογικές σκέψεις μαζί με το κείμενο, ακόμα και όταν αυτές αντιτίθενται στο ε, κείμενο ποτέ μετά από τόσα χρόνια στο Κοινοβούλιο δεν είδα μια τέτοια διαδικασία. Ε, στρέφουν το βλέμμα τους προς εμάς ε, όλοι οι εκπρόσωποι του κλάδου της ε, του πολιτισμού αλλά και οι ανταγωνιστές μας οι οποίοι μετρούν αυτή τη στιγμή την αδυναμία μας. Θα πρέπει για το θέμα αυτό να έχουμε ήρεμη ψηφοφορία και ορθή, σωστή ψηφοφορία. Αυτά ήθελα να πω εξ αρχής και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ε, για το ψηφιακό περιεχόμενο είχαμε μια τέτοια ε, ψηφοφορία αλλά και βάσει ε, του άρθρου 174 αποφάσισα να οργανώσω την ψηφοφορία με αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε να διευκολυνθεί. Αναφέρομαι στην σχέση μεταξύ αιτιολογικών σκέψεων και κειμένου αλλά κύριε Καβαδά Κύριε Καβαντά, εάν κατάλαβα καλά, ζητάτε να γίνει χωριστά η ψηφοφορία ο κύριος εγώ σας ζητώ να γίνει χωριστή ψηφοφορία για τις αιτιολογικές σκέψεις όταν το περιεχόμενό τους αντιτίθεται στο κείμενο. Όταν το περιεχόμενο των αιτιολογικών σκέψεων είναι ταυτόσιμο με αυτό του κειμένου δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά είναι απαράδεκτο κύριε Πρόεδρε όταν το περιεχόμενο της αιτιολογικής σκέψης αντιτίθεται στο περιεχόμενο του αρχικού κειμένου ε, τότε ε, ε, δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε τη δυνατότητα να ψηφίσουμε χωριστά. Γιατί, ε, εν πάση περιπτώσει, τότε να ψηφίσουμε unblock για όλο το κείμενο χωρίς καμία χωριστή ψηφοφορία. Πρόεδρος, ε, η γραμματεία μας είπε ότι δεν ε, ισχύει αυτό που λέτε, δηλαδή ότι αιτιολογικές σκέψεις έχουν διαφορετικό περιεχόμενο ή αντίθετο περιεχόμενο από τα άρθρα. Ο κύριος Καβαντά. Ναι, θα ήθελα να ζητήσω παρακαλώ από τη γραμματεία να διαβάσει προσεκτικά το κείμενο γιατί προφανώς δεν το έχει πράξει. Πρόεδρος. Παρ' όλα αυτά, και ε, για να σεβαστούμε το αίτημά σας ε, θα κάνουμε χωριστές ε, ψηφοφορίες. ο κ. Καβαδά, σας ευχαριστώ πολύ. Ήδη βελτιώθηκε η κατάσταση με αυτήν την πρότασή σας. Η κυρία Ρέντερ. Um, uh, Πρώτα, συζητήσαμε όλες τις αιτιολογικές σκέψεις που έχουν σχέση με μια συγκεκριμένη συμβαστική τροπολογία και έχουν συζητηθεί από κοινού και έχουν συμφωνηθεί από τις πολιτικές ομάδες. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος ψηφοφορίας επειδή εδώ υπάρχει κάποια διαφωνία. Κάθε πολιτική ομάδα έχει την ελευθερία να μην υπερψηφίσει εάν δεν ικανοποιείται από κάποιο στοιχείο. Δεν θα πρέπει όμως να μπορεί να ψηφίσει υπέρ ενός τμήματος της συμβαστικής τροπολογίας και κατά ενός άλλου. Επίσης θα ήθελα να αντιταχθώ στην τροπολογία του κ. Καρύμ για την τροπολογία 12, την προφορική τροπολογία για το άρθρο 11 του κ. Καβαντά και την προφορική τροπολογία του εισηγητού για τη συμβαστική τροπολογία 12 για την αιτιολογική σκέψη 33. Πολύ ευχαρίστω να κάνω τι παρατηρήσει αυτέ και στη διάρκεια τη προφορία. Αλλά ε, ε, εξ όσων έχω καταλάβει, εάν κανεί επιθυμεί να προβάλλει ένσταση κατά μια ε, προφορική τροπολογία, οφείλει να το πράξει ε, από την αρχή της ψηφοφορίας. Για ποιο λόγο ενίσταστε κυρία Σρέντερ. Ενίσταμε διότι είχαμε προθεσμία για την τελικοποίηση των συμβαστικών τροπολογιών, ώστε και οι άλλες πολιτικές ομάδες να έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν μια ημέρα αργότερα εναλλακτικέ τροπολογίες που να απηχούν ε, την έκβαση της συζητήσεως. Εάν μια συμβαστική τροπολογία τροποποιηθεί μετά από την κατάθεση των ε, εναλλακτικών ε, τροπολογιών, τότε η έκβαση γίνεται πολύ αβέβαια. Γι' αυτό και είμαι αντίθετη με αυτές τις τρεις τροπολογίες. Και το πρώτο αυτό εξ ονόματος της ομάδας μου Πράσινη EFA. What, what can I tell you? Uh, Πρόεδρος, και τι να σας πω τώρα. Θεωρώ ότι η ένσταση αυτή δεν έχει καλός. Διότι Because your, uh, your objection is... Διότι η ένστασή σας δεν συμβαδίζει με τους λόγους που προβλέπει ο κανονισμός. Μια στιγμή να κοιτάξω. Yes. Uh, uh, if you look at uh, Εξετάστε το άρθρο 169, παράγραφος 6. Μπορείτε να προβάλλετε ένσταση, για παράδειγμα, επειδή οι προφορικές τροπολογίες δεν ήταν διαθέσιμες σε κάποια από τις επίσημες γλώσσες εργασίας. Ιδάλλως, ο λόγος που επικαλείστε δεν είναι ορθός. Ο κύριος Βος. Σρέντερ, δεν γνωρίζω να έχουν ε, διανεμηθεί οι ε, προφορικές τροπολογίες σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Εσείς κύριε Φως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ε, που επιτρέπετε και στον εισηγητή να πει κάτι. Πρώτα λοιπόν σήμερα έχουμε φτάσει στο παρόν κείμενο μετά από πολλές και μακρές συνεδριάσεις. Έχουμε καταλήξει το κείμενο που έχουμε τώρα μπροστά μας. Ο χρόνος δεν ήταν περιορισμένος και γι' αυτό επιθυμώ να ευχαριστήσω όλες και όλους που συνέβαλαν στην προσπάθεια και βεβαίως και την γραμματεία η οποία εργάστηκε νύχθη για τη σύνταξη του καταλόγου ψηφοφοριών. Ε, δεν παίζουν ρόλο αυτά όμως, διότι θεωρώ ότι ως πολιτικές ομάδες θα πρέπει να σκεφτούμε και να συζητήσουμε και τα ουσιώδη θέματα έστω και, έχουν, αν έχουν περιβληθεί τρομανδία προφορικών τροπολογιών και να τα ψηφίσουμε επομένως. Θεωρώ ότι είναι υπερβολικά, είναι μάλλον τόσο σημαντικό το θέμα, ώστε δεν θα έπρεπε να γίνουν δεκτά διάφορα διαδικαστικά παιχνίδια. Για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε τώρα από το αδιέξοδο ανάμεσα σε μια ενδεχόμενη απόρριψη των προφορικών τροπολογιών, θα ζητήσω να αναβάλουμε την ψηφοφορία, ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε την όλη αυτή προσπάθεια σε μια διαδικασία που να είναι απολύτως στεγανή. Να μην μπορεί δηλαδή να προβληθεί καμία διαδικαστική ένσταση. Προτιμώ να ανοίξουμε και άλλη μια φορά λοιπόν την τροπολογία για εναλλακτικέ έστω τροπολογίες και να το συζητήσουμε και ψηφίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση. Διότι δεν έχει κανένα νόημα να πούμε τώρα ναι για τακτικούς λόγους για λόγους τακτική δηλαδή, ή να μην επιτρέψουμε κάτι για λόγους τακτική, προτιμώ να διεξαχθεί η ψηφοφορία σε έφθετο χρόνο επί των ουσιαστικών θεμάτων. Πρόεδρος, 190 παράγραφος 4. Επικαλούμε το άρθρο αυτό και θέτω την πρότασή σας ευθύς αμέσως σε ψηφοφορία. Όχι δεν μπορώ να δώσω το λόγο, πρέπει και οφείλω να δώσω να ε, θέσω σε ψηφοφορία αμέσως την πρόταση του εισηγητού για αναβολή της ψηφοφορίας. Και το πράττω αυτό ηλεκτρονικά. Η ψηφοφορία αρχίζει. Ένα πλεονάζον μέλος των, ε, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ένα μέλος παραπάνω, εξ όσων δικαιούστε. Άλλος ένας κύριε πρόεδρος. Μόνο 24 ψηφίζεται αυτή τη στιγμή. Καλώς. Κλείνω. Η πρόταση απερίφθη λοιπόν λόγω ισοψηφία. Η κυρία Γκέριγκερ ζητεί το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα ε, και πριν, είχα ζητήσει δηλαδή και πριν να πάρω το λόγο. Ε, ήθελα να σας πω ότι η εργασία μας σε περίπου δύο χρόνια και ε, η εργασία αυτή ε, ακριβώς περιλαμβάνεται στις συμβιβαστικές τροπολογίες τις οποίες από κοινού ε, έχουμε προωθήσει και χαίρομαι που προχωράμε με την ψηφοφορία σήμερα γιατί διαφορετικά θα είχαμε ακόμα μεγαλύτερο, πιο χαοτική κατάσταση, μεγαλύτερο χάος. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε. Ας ψηφίσουμε λοιπόν. That means that we go to the vote. Προχωρούμε στην ψηφοφορία, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Σρέντερ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επαναλάβω την ένστασή μας κατά των προφορικών τροπολογιών. Δεν πρόκειται για τεχνική λεπτομέρεια. Υπήρχε ψηφοφορία για... Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Υπήρχε προθεσμία για τι ε, προφορικέ τροπολογίε, Ορισμένα από τα κείμενα που προβάλλονται τώρα στις προφορικές τροπολογίες συζητήθηκαν στους σκιώδεις συζητητές και απερίφθησαν και μετά το πέρα τη προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών οι άλλε ομάδε είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν εναλλακτικέ τροπολογίε. Και όταν πέρασε η προθεσμία αυτή, οι αρχικέ συμβαστικές τροπολογίε αλλάζουν. Δεν μας μένει πλέον άλλη δυνατότητα να αλλάξουμε την θέση μας. Γι' αυτό και πρέπει να ψηφίσουμε τις αρχικές συμβαστικές τροπολογίες. Επιπροσθέτως, ως πρόσθετο επιχείρημα, δεν έχουν διανεμηθεί όλες οι προφορικές τροπολογίες σε όλες τις επίσημες γλώσσες, σε όλους τους ευρωβουλευτές. Εσείς, Κάουφμαν. κυρία Κάουφμαν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Προβλέπω η ψηφοφορία να διεξαχθεί αρκετά περίπλοκα. Προτείνω λοιπόν να γίνουν όλες οι ψηφοφορίες, όλη η ψηφοφορία δηλαδή να γίνει ηλεκτρονικά. Ο πρόεδρος, θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά η ψηφοφορία, θα γίνουν ψηφοφορίες κατά τμήματα, όπως ζήτησε ο κ. Καβαντά, και οι προφορικές τροπολογίες που δεν συνδέονται με τις συμβιβαστικέ που θα ψηφιστούν πρώτες. Οι προφορικές τροπολογίες μπορούν να ψηφιστούν και στη διάρκεια της διαδικασίας ψηφοφορίας. Right. So we Ας αρχίσουμε. Ορίστε. Σρέντερ. Σύμφωνα με το άρθρο 170, το οποίο εφαρμόζεται στις ψηφοφορίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπές, δύο μέλη της Επιτροπής έχουν το δικαίωμα να προβάλλουν ένσταση σε προφορική τροπολογία η οποία ε, τίθεται ψηφοφορία. Και αυτό πράττουμε. Θα αποφασίσουμε τότε επί των επιμέρους ενστάσεων όταν θα φτάσουμε στην ψηφοφορία. Κυρία Γκέριγκερ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε κύριε Πρόεδρε την ψηφοφορία και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε παρακαλώ τον κατάλογο για την ψηφοφορία όπως έχει διατυπωθεί οι συζητήσεις που έγιναν μέχρι τώρα και οδήγησαν στον κατάλογο αυτό ε, περιελάμβαναν και τα συγκεκριμένα άρθρα και τις αιτιολογικές σκέψεις. Τώρα το να ψηφίσουμε ε, με ξεχωριστό τρόπο πράγματα τα οποία συζητήθηκαν από κοινού είναι λάθος. Οι συζητήσεις, επαναλαμβάνω, έγιναν από κοινού ανάμεσα ε, ε, σε αιτιολογικές σκέψεις και σε αρχικό κείμενο. Συνεπώς έτσι θα πρέπει να προχωρήσουμε, έτσι έχει διατυπωθεί, έτσι έχει συνταχθεί ο κατάλογος ψηφοφορίας. Αν υπάρχουν τέτοιες αντιρρήσεις θα μπορούσαμε να τις είχαμε συζητήσει νωρίτερα και θα μπορούσαμε να κάνουμε την ξεχωριστή ψηφοφορία. Όμως τώρα τα πράγματα έχουν ε, πλέον διαμορφωθεί και θα πρέπει να παραμείνουν ως έχουν. Πρόεδρος, κύριε Γκέριγκερ, δυστυχώς δεν μπορώ να δεχτώ την αίτησή σας και επικαλούμε το άρθρο 174 παράγραφος 7. Εάν μια πολιτική ομάδα και υποθέτω ο κ. Καβαντά μιλούσε εξ ονόματο της Άλντε. Εάν ζητήσει η ψηφοφορία κατά τμήματα, τότε η ψηφοφορία κατά τμήματα οφείλει να διεξαχθεί. Καλώ. Συνεχίζει ο πρόεδρος. Αρχίζει η ψηφοφορία. Αποφασίσαμε λοιπόν να την διεξαγάγουμε καθ' ολοκληρία ηλεκτρονικά. Συμβαστική 1 και 1α. 1 bis. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα συγκρίνεται. Τροπολογία 497. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 498 αρχίζει εγκρίνεται. Πεντακόσια και πεντακόσια ένα. απορρίπτονται. Σαράτα ένα. Επιτροπής Πολιτισμού. Θα απλουστεύσω κάπως την διαδικασία, δεν θα επαναλαμβάνω διαρκώς την φράση ότι αρχίζει η ψηφοφορία ή ότι λύγει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται λοιπόν η 41. 506 και 507. Απορρίπτονται. 508. Εγκρίνεται. 504. απορρίπτεται. Ήμκο 34. Απορρίπτεται. 509. Απορρίπτεται. 510. απορρίπτεται. 511 εγκρίνεται. Τροπολογία 30.

απορρίπτεται 29 πέρας απορρίπτεται 514 πλεονάζει μια ψήφος του Λαϊκού Κόμματος. Απορρίπτεται λοιπόν 514, 515, Απορρίπτεται. 42. απορρίπτεται 36 απορρίπτεται συμβιβαστική 3 εγκρίνεται 516 τροπολογία. 516 δεκαέξι επαναλαμβάνει ο Απορρίπτεται. 517 απορρίπτεται. Ήμκο 37. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 20α, 20 bis. απορρίπτεται. Συμβιβαστική 20. Εγκρίνεται. Τροπολογία 524. Απορρίπτεται. 425. Απορρίπτεται. Ήτρε 34. Απορρίπτεται και αυτή. 526. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Εγκρίνεται.

εγκρίνεται. Τροπολογία 567. Άρθρο 3. Α νέο. Πρόκειται για την 567 τροπολογία που αφορά το άρθρο 3α νέων. Απερίφθη. Συμβαστική τροπολογία 5. εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Στη σελίδα 15 της λίστας και πρόκειται για το άρθρο 5. Συμβαστική 7. Σελίδα 14 στο έγγραφο. Εγκρίνεται. Συμβαστική 58. αφορά το άρθρο 5α νέο. Ξαναλέει ο πρόεδρος, συμβαστική τροπολογία 58. Κλείστε την ψηφοφορία παρακαλώ. Αυτή απερίφθη λοιπόν. Τώρα λοιπόν η τροπολογία 658. Ακριβώς από κάτω. Απερίφθη. 659 και ΙΜΚΟ 55. απορρίπτονται. 869 απορρίπτεται. 871. Α, συγγνώμη, 871. 871. Απερίφθη.

απορρίπτεται 662 απορρίπτεται και αυτή 663 απορρίπτεται συμβιβαστική 56

απορρίπτεται 666 απορρίπτεται 667 μαζί με την ΙΜΚΟ 54 απορρίπτονται 668. Απορρίπτεται. 669. Απορρίπτεται. 670. απορρίπτεται 671 απορρίπτεται ΙΜΚΟ 56 απορρίπτεται Τροπολογία 672. Εγκρίνεται. 674. Απορρίπτεται. 675. απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Μια στιγμή να δούμε και πού βρίσκεται. Συμβαστική 9 ψηφίζεται για τη συμβαστική 9 που αφορά το άρθρο 8. Εγκρίνεται συμβαστική 10 επί του άρθρου 9. Εγκρίνεται. Τροπολογία 722. Απορρίπτεται αυτή. Συμβιβαστική τροπολογία 11. Εγκρίνεται ανθρωπολογία 728. Απορρίπτεται. 51. εγκρίνεται.

απορρίπτεται. Κυρία Σέντερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα τώρα να προβάλλω ένσταση επί της προφορικής τροπολογίας του κυρίου Καρίμ και του κυρίου Καβαντά. Αντιλαμβάνομαι ότι και οι δύο θα προσθεθούν στην ε, συμβαστική τροπολογία 12. Και εάν ερμηνεύω σωστά το άρθρο 209, ζητώ την υποστήριξη ενός ακόμη μέλους. Αλλά δεν χρειάζεται να γίνει εξ ονόματος, μάλλον προβάλλω αυτή την αίσθηση εξ ονόματος της ομάδας των Πρασίνων EFA.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 Α, είναι τρεις συνολικά. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Ο κύριος Καβαντά. Εγώ θα ήθελα να υποβάλω την τροπολογία μου, έστω και αν υπάρχει αντίθεση. Ναι, τροπολογία για το 11. Très bien. Uh, Ο Πρόεδρος. Θα ψηφίσουμε τώρα την συμβιβαστική τροπολογία 12 χωρίς την προφορική τροπολογία. Αυτό θα ψηφίσουμε τώρα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Μπορείτε να ανοίξετε παρακαλώ την ψηφοφορία. Δεν τίθεται το θέμα λοιπόν των προφορικών τροπολογιών μετά από την ε, ψηφοφορία αυτή και προχωρούμε. Η κυρία Σρέντερ, υπάρχει ακόμα μία προφορική τροπολογία επί των αιτιολογικών σκέψεων. προχωρούμε με την ψηφοφορία για την τροπολογία 785. ...785 που αφορά το άρθρο 11α νέο.

γραμματεια του Συμβαστική Τροπολογία 14Β. Απερίφθη. Ήμκο 67 και Λίμπε 7. εγκρίνεται.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 εγκρίνεται. 8.72 απερίφθη. Κάλτ 86 εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15α, 15 bis. Απερίφθη. Συμβιβαστική 15β, 15 ter. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16